Όπω όπως προβλέπει ο κανονισμός. Από την πολιτική ομάδα ΑΛΔΕ έχουμε ε, λάβει την εξανακοίνωση η κυρία Πατσιαλαλών ως ε, τακτικό μέλος θα συμμετάσχει στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ο κύριος Κυρί Κορνιγέ ως τακτικό μέλος της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων και Νομισματικών Υποθέσεων. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση, οι ορισμοί αυτοί θα